Uh, dear friends, ladies and... Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, 60 δευτερόλεπτα μέχρι την έναρξη της συνεδρίασής μας. Σας παρακαλώ καθίστε. Διότι θα ξεκινήσουμε αμέσως, τώρα. All of you, advisors as well. Advisors from the EPP group as well. Great. Τέλεια. Καθίσαμε και ε, του ΕΛΚ και όλοι οι άλλοι από το ECR. Okay. <laughs> okay, sorry. Sorry, sorry. Dear friends. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα παρακαλώ ησυχία, γιατί διότι έχω πολύ σημαντικές πληροφορίες να σας δώσω. Μ' ακούτε όλοι? Ωραία. Σήμερα στη μία θα ξεκινήσουμε την, ολομέλεια, την κοινοβουλευτική ολομέλεια της ενεργειακής κοινότητας. Οι συνάδελφοί μας από τα Δυτικά Βαλκάνια, έξι χώρες, καθώς και Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία, θέλουν να συναντηθούν μαζί μας. Την προηγούμενη φορά ταξίδευσαν χιλιάδες χιλιόμετρα και τελικά μόνο δύο ευρωβουλευτές ήταν παρόντες. Έχουμε αρκετού αδέρφους και από τις ανατολικές χώρες ε, και σχεδόν ε, κανένας ε, ευρω... από την Ήτρε δεν ήταν παρόν. Και είναι ντροπή αυτό διότι το 2005 ξεκινήσαμε με βάση πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εννέα χώρες γειτονικέ μας προσπαθούν να υιοθετήσουν του ίδιους κανόνες που εφαρμόζουμε και εμείς. Έχουμε λοιπόν μια ενεργειακή ένωση 36 ε, χωρών. Σας παρακαλώ ελάτε έστω και για ένα τέταρτο, για 20 λεπτά. Πριν την συνάντηση θα σερβίρουμε ε, ένα μικρό γεύμα, μπορείτε να έρθετε στη μία η ώρα δηλαδή, για να φάτε κάτι ελαφρύ. Δεν χρειάζεται δηλαδή καν να πάτε για φαΐ. Ακόμα λοιπόν και για 20-25 ε, λεπτά, μισή ώρα παρακαλώ να έρθετε. Και στις 2.30 ξεκινάει η συνεδρίαση της Ήτρε. Αυτά λοιπόν, μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Παρακαλώ. Πατήστε το κουμπάκι. Δεν βλέπω αρκετούς συναδέλφους να έχουν ψηφίσει. 52. Μα τι, δεν είναι κανείς παρόν. Δεν λειτουργεί. Ah, mine, mine is not working. Φαίνεται να μην λειτουργεί η δική μου συσκευή. What is going on? Oh, no. Okay. Okay. Uh, thank uh, Λήξη της, ε, ψηφοφορίας. It's draft opinion. Σχέδιο έκθεσης που καθιερώνει πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ράινχαρτ Μπιουτικόφερ είναι ε, συντάκτη ε, τη νομοδότησης, ε, συμβιβαστική 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ένα τέσσερα τρία Χωριστή ψηφοφορία ζητάει η Γκουε. περιβαλλοντικά πρότυπα ε, υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Rejected. Uh, απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση της 16, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 149 υπέρ. 149 υπέρ. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2D ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 164. And I close the vote. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Yes, of course. Uh, it's um, amendment Τροπολογία 165. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική 2C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3d υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3e υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. 192. Παρακαλώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν ψηφίσαμε το δεύτερο τμήμα της 185. Ναι, έχετε δίκιο. amendment Τροπολογία 185, το δεύτερο τμήμα. Επειδή είναι γκρίζο, αλλά έχετε δίκιο. Πρέπει να το ψηφίσουμε. Πάμε πίσω λοιπόν πριν την 3α, 185 δεύτερο τμήμα και ζητώ συγγνώμη. Πρόκειται για δική περίπτωση. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας αυτής. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3 ή. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3F υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 208 κατά τα ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, το πρώτο τμήμα. 208, το πρώτο τμήμα. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται και πάλι. Ναι, φυσικά λέει ο πρόεδρος. Part two. Το δεύτερο τμήμα, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική απαλήθευση δεν είναι πολύ σαφής κατάσταση 24. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 και 2.32 είναι πανομοιότητες. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 233 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 ε, ε, υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. 30. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, την 271 ελέγχουμε λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 7α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. 42. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 7D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, ευχαρίστως λέει ο πρόεδρος ηλεκτρονική επαλήθευση. 306, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 8α, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8β, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 322 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 321 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 330 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 59. I Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 ηλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Α, ηλεκτρονική απαλήθευση. 66 η ηλεκτρονική επαλήθευση της 66. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 67 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 68 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 69 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 70 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της 73 I close the vote. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται 74 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 74. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 74, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, 75 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της 85. And I close the vote.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 98 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 98. I close the vote. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση και πάλι. Για να είμαστε βέβαιοι. I close the vote. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 8. And I close the vote. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. 133. And I close the Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία πάνω στο σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία φυσικά. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τελειώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες ε, για την ε, έκθεση αυτή. Στη συνέχεια έχουμε το θέμα της ελεύθερης ροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κράσνοντέψκι είναι συγητής, συμβαστική 1, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά για να ελέγξουμε την 63 λήξη απορρίπτεται 64 υπέρ κατά να ελέγξουμε 64 ελέγχουμε την τροπολογία 64 πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 33. Λήξη της ψηφορίας. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε και πάλι την 35. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. 41. Και λήξη της ψηφοφορίας. Δεν γίνεται αποδεκτή αυτή τη φορά. 42 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε τη 43. Πέρας. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Έχουμε συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον συγητή. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σχέδιο γνωμοδότησης. Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή. Η κυρία Ματία είναι η 35 υπέρ κατά αποχές Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μήπως ε, θα πρέπει να σε μπλοκ όχι 53 υπέρ κατά 53 για να την ελέγξουμε την 53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 κατά εποχές εγκρίνεται, συμβαστική 1 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ, κατά εποχές απορρίπτεται, συμβαστική 3 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται, συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 30 υπέρ,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 Λοιπόν, γλωσσική το Μαρίσα Σαματίας, λήξη της πληροφορία, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα περνάμε στους κανόνες και γενικές ε, αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη-μέλη και των εκτικών διασμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, με συγχωρείτε. Λοιπόν, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά για να ελέγξουμε συμβαστική 2 λήξη εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά για να ελέγξουμε. Συμβαστική 4. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε αυτή τη συμβιβαστική τροπολογία. Πιθανότατα θα γίνει αποδεκτή. Λήξη. Εγκρίνεται. Βεβαίω. Πάμε τώρα στο 18. Υπέρ. Κατά. Για να ψηφίσουμε, γιατί δεν είναι σαφές, να ψηφίσουμε για τη 18. και την 7 μαζί. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Είχαμε κοινή ψηφοφορία με την 7. Γιατί και δύο πρέπει να ψηφιστούν μαζί. 47 υπέρ. Κατά εποχές, να το ελέγξουμε για τις 47. Λήξη. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε τη 19. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε και την 20. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί δεν μπορώ να βλέπω. Λήξη της πληροφορία για την τροπολογία 20 εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε τη συμβιβαστική 6. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 και 8 μαζί. Υπέρ. Κατά για να ελέγξουμε. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά ας το δούμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία και τώρα λήξη της ψηφοφορίας. Λοιπόν, ε, άσκηση εκπληστικών αρμοδιοτήτων.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 Thank Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. our rapporteur, uh, colleague Jens Geyer, is not. Δεν είναι εδώ η μου, ο Γιάννης Γκάιερ, και γι' αυτό θα πρέπει να τον περιμένουμε. Από την άλλη, βέβαια, ο Γενικός Εισηγητής για τον Προπολογισμό του 2019, ο Ντανιέλε Μπιόνκι είναι εδώ μαζί μας αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τον εισηγητή μας τον Γιέντς Γκάιερ σε ένα λεπτό θα είναι μαζί μας από όσο ξέρουμε yeah. Uh, Paul Rubik, κύριος Ρούμπεκ υπό τα διάφορα. Καλή ιδέα. Να δούμε τώρα κάτι που είναι υπό τα διάφορα. Ναι, ήθελα να, να θυμίσω ότι στις 17 Μαΐου θα είναι εδώ ο Επίτροπος Μοήρας και έχουμε λάβει, λάβει και την απάντηση για το Κιώτο στην Ιαπωνία θα ζητήσω από τους συναδέλφους στις 17 Μαΐου το απόγευμα που θα γίνει μια συζήτηση για την ανοιχτή επιστήμη Open Science και Global Competition. Ε, θα έχουμε και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε περίπου τρεις σελίδες για το FP9 εκεί. Στις 17 ε, Μαΐου λοιπόν θα είναι εδώ ο κ. Μοέιρας ε, και θα είναι χρήσιμο εκείνη τη μέρα να ξεκινήσει η διαδικασία fast track να σκεφτούμε λοιπόν ε, κάποια στρατηγική έτσι ώστε ως εκείνη τη μέρα να είναι σαφές το Κοινοβούλιο ε, δίνει τη μάχη ε, για το FP9 να εγκριθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα δηλαδή. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω τον Πασκάλ Λαμή για τον διπλασιασμό του προπολογισμού. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν 17 Μαΐου έτσι ώστε η Ήτρε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ. Όντως, ε, την 5η 17 Μαΐου έχουμε αυτή την παρουσίαση του FP9 με ιδιαίτερη επικέντρωση στη διεθνή συνεργασία ο συνάδελφος Ρούμπι, ο κ. Μόντερς ε, καθώς και οι Ιάπωνες εκπρόσωποι θα είναι εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ που μας το θυμήσατε. Λοιπόν, ο Γιάννης Κάιερ είναι εδώ μαζί μας, μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ανταλλαγή απόψεων για τον προπολογισμό του 2019 με τον Ντανιέλ Μπιόντι, ο οποίος είναι ο εισηγητής της Επιτροπής Προπολογισμού. Ο δικό μας ε, ε, ε, εισηγητής είναι ο κύριος Γκάιερ της Επιτροπής Ήτρε η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τον προβλησμό στο τέλη Μαΐου ως το συνήθως η γνωστή διαδικασία είναι μικρός, ο, μικρό χρονικό διάστημα από την δημοσίευση ως τη συζήτηση τον Ιούνιο μπορούμε λοιπόν να δώσουμε τη γνώμη μας για την εντολή σχετικά με τον Τρίλογο υπό τη μορφή επιστολής και αυτό συνηθίζεται πάντως γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να ε, επεξεργαστούμε αυτήν την ειδική νομοδότηση. Θέλουμε πάντως επιστολή στην Δημοσιονομική Επιτροπή. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 10 Ιουλίου για τις δημοσιονομικές γραμμές Ήτρε και το ψήφισμα 24 Σεπτεμβρίου ε, Βεβαίως όλοι καλείστε να υποβάλλετε ιδέες για τα προγράμματα ε, στείλαν τες ε, στην Επιτροπή, στην Συγγραμματεία της Ήτρε έως 24, Απριλίου το αργότερο, δηλαδή σήμερα. Έχουμε λοιπόν χρόνο για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που είστε εδώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ανημερώσω τα μέλη ότι πρώτα απ' όλα θα μιλήσει ο συνάδελφος ο κύριος Μπιόντι, ο εισηγητής και στη συνέχεια ο κύριος Γκάιερ. με φίλε από την Δημοσιονομική Επιτροπή έχετε το λόγο. Κύριε Βιώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ και την Επιτροπή που θέλησε να με ακούσει και τώρα θα επικεντρωθώ σε ορισμένα σημαντικά σημεία. Όμως, ε, εν τω μεταξύ, θέλω να αναφερθώ και στην ε, διαδικαστικά. Σκοπεύω να συνεργαστώ με όλες τις επιτροπές και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έχουμε όσο το δυνατόν ε, μία εντολή και μία πρόταση για τον προϋπολογισμό που να την χάνουν ε, τις μεγαλύτερες συνένεσεις από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Να είμαστε λοιπόν ισχυροί τη στιγμή που θα πάμε στη συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο. Και στρέφομαι κυρίως στη δική σας Επιτροπή που έχει ένα θεμελιώδη ρόλο να διαδραματίσει. στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι σίγουρα θα έχετε διαβάσει το έγγραφο ε, που ψηφίσαμε, τις κατευθυντήριες γραμμές του προπολογισμού που ψηφίσαμε το Μάρτιο στην Ολομέλεια και θα έχετε δει πως ε, η σημασία θέλουμε να δώσουμε στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή Ήτρε. Θα τα αναφέρω πολύ σύντομα για να κατανοήσω αν συμφωνούμε στις προτεραιότητες και στη συνέχεια θα ακούσω τις δικές σας προτεραιότητες. Θα ακούσω δηλαδή την τοποθέτηση του κυρίου Γκάιρ με τον οποίο συνεργαζόμαστε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Φυσικά αυτό θα διευκολύνει και το έργο της δικής σας Επιτροπής ε, και τη συνεργασία με την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Καταρχήν, εμείς ε, πρέπει να εφαρμόσουμε του στο 1 1α και τη χρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων ορίζοντας 2020 κόσμε και ε, κυρίως στον ορίζοντα 2020 πρέπει να εγγυηθούμε ότι έχουμε το κατάλληλο επίπεδο κονδυλίων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για να ενισχύσουμε την έρευνα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες την Ευρώπη σε έναν κόσμο που αλλάζει ε, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινδύνου και το μηχανισμό για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Εντός ε, της χρηματοδότησης του κόσμου ε, τα κονδύλια θα πρέπει να αυξηθούν. Έχουμε και διατάξεις για τις ΜΜΕ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ευνοϊκό κλίμα για την επιχειρηματικότητα και να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους ερευνητές ε, και επιχειρηματίες να ξεκινήσουν ε, τις δικές τους πρωτοβουλίες. Εμεί ε, θέλουμε να έχουμε χρηματοδότηση για τα ΕΦΗ e e δίκτυα, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την καταπολέμηση των εκπομπών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καταπολέμηση κατά της ενεργειακής ανέχειας θα πρέπει ε, να προωθήσουμε αυτό το στόχο, να έχουμε τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να αναστρέψουμε τις περικοπές που προβλέπονται για τον ορίζοντα 2020 και για το πρόγραμμα ε, MCE. Ε, να εγγυηθούμε τουλάχιστον το 20% του προπολογισμού της Ένωσης ε, θα ξοδεύεται για δράσεις για το κλίμα και για τη μείωση των εκπομπών άνθρακαν. Αυτά τα δύο σημεία είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά από τη δική μας σκοπιά. Η χρηματοδότηση του προγράμματος ανάπτυξης επίσης και στον τομέα της άμυνας είναι σημαντικό. Πρέπει να εγγυηθούμε ότι η ανάπτυξη αυτού του νέου προγράμματος να μην οδηγήσει στην αφαίρεση πόρων από υφιστάμενα προγράμματα. Αλλά η αρχή που μας ε, καθοδηγεί είναι ότι θα πρέπει να έχουμε νέα χρηματοδότηση για αυτό το πρόγραμμα για τον τομέα της άμυνας. πρέπει να υπάρχει η εγγύηση ότι θα τρέξουν μακροπρόθεσμα τα προγράμματα, πρέπει το Κοινοβούλιο να αναλάβει μια δέσμευση απέναντι στους ερευνητές, απέναντι στους πολίτες. Επίσης πρέπει να αποφύγουμε τις περικοπές και να δώσουμε ένα χρηματοδότηση για τους οργανισμούς ε, της Ένωσης προκειμένου να μπορούν να αναλάβουν νέα καθήκοντα. Φυσικά έχω κατά νου την περίπτωση της ΕΝΗΣΑ. Αυτά είναι τα κύρια θέματα επιτάπητος. Ε, βέβαια είμαι εδώ για να ακούσω και εσάς και να πάρω σημειώσεις προκειμένου να μπορέσω να αυξήσω ε, τις πληροφορίες που θα έχω στη διάθεσή μου. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο εισηγητής μας, ε, ο Γιάννης Γκάιερ, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι τα πράγματα έχουν όπως τα περιέγραψε ο Τανιέλε, διότι είμαστε ε, και οι δύο μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού και έτσι παίζουμε πινκ-πονγκ μεταξύ μας. όσον αφορά τις ειδικέ ανάγκες της Επιτροπής Ήτρε. Σας ε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Ε, πάντως ε, ασχολούμουν με το θέμα αυτό, διότι στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, στο κτίριο Γιάν, δηλαδή αρκετά μακριά από τη δική μας αίθουσα, συζητούσαμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με έναν ε, συμπληρωματικό προϋπολογισμό, διορθωτικό προϋπολογισμό για τους πρόσφυγες ε, στο, στην Τουρκία. και προσπαθούσαμε να συμφωνήσουμε σχετικά με την πληρωμή της δεύτερης δόσης, ε, δηλαδή ε, άλλα 3 ε, εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πολλές ε, δυνατότητες δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει πολλές δυνατότητες χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Το θέμα είναι να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη με έναν τρόπο όχι ιδιαίτερα επιβραντικό για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, κάτι που φαίνεται να αποτελεί απειλή αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να πω το εξή. Ο Ντανιέλ και εγώ ασχολούμαστε πολύ με την ε, πολιτική, τη δημοσιονομική πολιτική. Και μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού ε, έχει ήδη αποφασιστεί είτε όσον αφορά την ε, γεωργική πολιτική όπου οι γεωργοί έχουν ε, αξιώσει και είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε περικοπές ε, ή έχουμε την περιφερειακή πολιτική και τους εθνικούς φακέλους ε, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων ε, στις πολι... πολιτισμικές οικονομικές προοπτικές. Τι απομένει λοιπόν οι πόροι στους οποίους έχει πρόσβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ο ορίζον 2020 και η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Εάν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ανακατονομή των πόρων, τότε ε, αυτές τις δύο δυνατότητες έχουμε και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε στενά με τον ε, εισηγητή, διότι ο συνάδελφος Βιώτη έχει απόλυτο δίκιο. Ε, μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση μόνο εφόσον συμφωνούμε μεταξύ μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει δηλαδή να συμφωνήσουμε πέρα από τα όρια των πολιτικών μας ομάδων. Ε, στην Επιτροπή Προπολογισμού ε, συχνά υπάρχουν μεγάλες διαφορές απόψεων. Στηρίζουμε πάντως τις κατευθυντήριες γραμμές του συναδέλφου Βιώτη, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρξουν περικοπές στο ορίζον 2020, μάλλον θα πρέπει να ενισχυθεί το πρόγραμμα. Εμείς ε, με τρόμο διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μόνο κάθε έβδομο ε, επιτυχημένο ερευνητικό πρόγραμμα. Διότι ναι, είναι αρκετά μεγάλο το ορίζον 2020 σε σχέση με τον γενικό ε, Παρ' παρόλα αυτά συνεχίζει να μην αρκεί. Δηλαδή θα μπορούσαμε τα εφταπλάσια προγράμματα να χρηματοδοτήσουμε αν είχαμε επαρκείς πόρους. Η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα θα μπορούσαν έτσι να ενισχυθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν αύξηση και όχι μείωση. Χρειαζόμαστε αύξηση στο πλαίσιο του ορίζον 2020. για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα υπόλοιπα προγράμματα του ορίζουν 2020 αλλά και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή έτσι έχει η κατάσταση αγαπητοί συνάδελφοι δεν θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι του Συμβουλίου που λέει ότι θέλουμε την έρευνα στην άμυνα, επειδή όμως ε, τα κράτη-μέλη, επειδή κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτό δεν, ε, ε, δεν μπορούμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για αυτά, ας πάρουμε τα χρήματα από το ορίζον 2020. Θα πρέπει λοιπόν, και συμφωνούμε με τον συνάδελφο Βιώτη, αν το Συμβούλιο θέλει περισσότερα χρήματα για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, τότε θα πρέπει η χρηματοδότηση να προέρχεται από επιπλέον πόρους. Το να ε, ενισχύσουμε αυτήν την έρευνα εις βάρος όλων των άλλων προγραμμάτων του Horizon 2020, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος προσέγγιση, διότι θέλουμε περισσότερα ευρωπαϊκά αγαθά που να, ε, που να προωθούνται και να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι λιγότερα. Δεν μπορούμε λοιπόν απλά να κάνουμε ανακατανομή ε, του προϋπολογισμού που έχει ε, καθιερωθεί απλά για να έχουμε μηδενικό άθροισμα. Και το ίδιο ισχύει για τους οργανισμούς. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να εφαρμόζεται τελικά επί τόπου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας φορέας που να εναρμονίζει τα ευρωπαϊκά συστήματα. Και αυτό ακριβώς κάνουν οι οργανισμοί. Έχουμε δει την κατάσταση κατά το προηγούμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ο προϋπολογισμός ε, των θεσμικών οργάνων ε, να μειωθεί κατά 5%. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε περικοπές κατά 5% στο προσωπικό κάθε οργανισμού. και μόνο με ακατανομή μπορούσαν ε, να αυξήσουν οι οργανισμοί το προσωπικό τους, το οποίο σημαίνει δηλαδή μείωση σε άλλους οργανισμούς. Ε, συνάδελφοι, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού είμαι ο μόνιμος, επιτροπός, ε, είμαι ο εισηγητής για τους ε, οργανισμούς. Ε, και οι οργανισμοί μου λένε ότι έχουμε φτάσει στα όρια όσον αφορά τη μείωση του προσωπικού. Εμείς ε, λοιπόν μαζί με τα κράτη-μέλη όσον αφορά συγκεκριμένους ε, οργανισμούς όπως είναι ο Frontex για παράδειγμα θα πρέπει να φροντίσουμε να αυξήσουμε το προσωπικό τους. Η μείωση λοιπόν, η περαιτέρω μείωση του προσωπικού των οργανισμών ε, αποτελεί μεγάλη αυταπάτη, ωστόσο το Συμβούλιο εμένει σε αυτό. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε τους τομείς για τους οποίους είναι αρμόδια η Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Περνάμε στους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Σαλίνη. Ευχαριστώ. Οι εισαγωγικέ παρατηρήσεις των συναδέλφων ε, είναι εξαντλητικέ και ξεκάθαρες. Έχω βέβαια ένα σχόλιο ότι οι ελλείψεις που έχουν προκύψει από την ε, έλλειψη ύπαρξης πραγματικών ε, περιθωρίων οδηγεί στο να μην υπάρχει δυνατή παρέμβαση. Του τομείς που μπορούμε να παρεύουμε, εμείς έχουμε δύο κυρίες προκλήσεις, ε, το θέμα της ποσότητας και τους κανόνες. Το είδαμε και στον τομέα που αφορούσε τη Γεωργία, στο ποιο είναι το κομμάτι του προπολογισμού που καταλαμβάνει. Και βέβαια και οι κανόνες είναι σημαντικοί το αν θα υπάρχει νέος επαναπροσδιορισμός του προγράμματος ή όχι. Αυτό αφορά τον ορίζοντα 2020 και είναι ζωτικό το θέμα της καινοτομίας και της έρευνας. Επομένως, η πρόκληση για μας θα είναι να εγγυθούμε επαρκείς πόρους και να προσδιορίσουμε κανόνες που να επιτρέπουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ποιότητά της και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις και γύρω και μεσέ επιχειρήσεις να κρατηθούν ζωντανές και να μπορούν να καινοτομήσουν. Η καρδιά ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την κοινοτομία αποτελείται από τι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει. Έτσι, μια σοβαρή πολιτική προϋπολογισμού, ο πρώτος ε, στόχος που θα έχει είναι να είναι φίλοι των επιχειρηματιών. Ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα εργαλείο κοινωνική ε, πρόνοιας, είναι ένα εργαλείο που έχει δημιουργηθεί για να εγγυηθεί χώρο και ενέργεια σε όποιον ξέρει να παράγει αξία. Έτσι, από εκεί περνά και η δυνατότητα να έχουμε τους κατάλληλους πόρους για ένα επαρκές σύστημα πρόνοιας για τους πολίτες. Το ίδιο ισχύει και για το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη. Είδαμε την ε, κρίσιμη σχέση μεταξύ της μορφής μηχανισμού, όπως ο μηχανισμός συνδέοντας στην Ευρώπη, ε, που χρηματοδοτούν πολύ σημαντικές επενδύσεις στην ε, υποδομή και του ΕΕΦΣΗ εντό του σχεδίου Juncker. Υπάρχουν κάποιε επενδύσει που μπορούν να υποστηριχθούν από το ΣΕΦ, ενώ από το ΕΦΣΙ όχι. Παραδείγματο χάρη, είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα των ε, κρίσιμων υποδομών. Για τα, κατά τα λοιπά, πιστεύω ότι η δουλειά που θα κάνουμε, αν βασιστεί σε τέτοια εύρωστα κριτήρια, θα μπορέσει να ευνοήσει τη συνεργασία στην οποία αναφέρθηκαν οι δύο συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ για την παρατηρήση. Μέρος του Άλντε, κύριος Ρουκέπ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά ήδη έχουν λεχθεί. Δεν έχω κάτι καινούριο να πω. Αυτό που είναι προφανές είναι ότι σε ένα προπολογισμό που πάντα ήταν έτσι σφιχτός, η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησαν να δημιουργήσουν ειδικά προγράμματα, ειδικά κονδύλια για τα πιο σημαντικά ζητήματα για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτά ε, και στα πλαίσια του προπολογισμού των κρατών μελών και στα πλαίσια του γενικού προπολογισμού. Έτσι δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020, ε, το FP9, το πρόγραμμα Collecting Europe Facilities ε, και, ε, ε, και εδώ μπαίνουν και άλλε δραστηριότητε όπω η διαστημική ε, Ευρώπη. Εδώ δεν μπορούσαμε να βρούμε κρίσιμη μάζα από το κρατομελών ε, και δυστυχώς ε, τα κράτη-μέλη είναι αυτά που αποφασίζουν για τις ανάγκες του προπολογισμού και τέτοια προγράμματα. Το είδαμε αυτό κατά τη δημιουργία του Ταμείου Juncker, παραδείγματος χάρη, όπου μέρος του Ταμείου Εγγυήσεων πήγαμε και πήραμε τα χρήματα από προγράμματα που ήταν κεφαλαίων του σημασίας ε, συμφωνώ με αυτό που είπε και ο εισηγητή μας και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού. Ε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε ε, να έρχονται και να ε, πετσοκόβουν ε, ευρωπαϊκά κονδύλια, ευρωπαϊκό προπολογισμό ε, εκεί όπου μιλάμε για κεφαλαιώδη, τομεί τομείς όπως τον τομέα της έρευνας παραδείγματος χάρη πρέπει οπωσδήποτε να, να στηρίξουμε τις επενδύσεις τις παραγωγικές. Και οι παραγωγικές επενδύσεις είναι η ανάπτυξη, είναι η έρευνα, ε, είναι οι ε, ε, επενδύσεις της υποδομές ενέργειας και μεταφορών μέσω του, του Trading Euro Facilities. Είπαμε, είδαμε λοιπόν με πόσο ενθουσιασμό αυξάνεται ε, αυξάνονται οι αρμοδιότητε και τα προγράμματα των υπηρεσιών και με πόσο ενθουσιασμό επίση πετσοκόβουν τον προπολογισμό του. Ε, και αυτό είναι ένα παράδοξο. Ο προπολογισμό του 2019 ε, παρουσιάζει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, διότι δίνει στην, ε, στο κοινοβούλιο μα τη δυνατότητα να δείξει την αποφασιστικότητά του και εν ώψη θα συζητήσεων για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Κοινοβούλιο δηλαδή πρέπει ξανά και ξανά να λέει ότι η προσθέμενη αξία η ευρωπαϊκή είναι αυτό το, είναι το κύριο μέλημα του προπολογισμού. Και, και για τη συζήτηση για τον προπολογισμό και για τη συζήτηση για το δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, σύντομα θα έχουμε και τι προτάσει τη Κομισιόν σχετικέ, ε, είναι απαραίτητο εμείς σε πολιτικό επίπεδο να επαναλάβουμε τις προτεραιότητε μα, να επαναλάβουμε ε, τι είναι αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε, αλλά και τι αρνούμαστε, ε, τι δεν δεχόμαστε. Ε, βλέπουμε για το πρόγραμμα σχετικά με τις αντισταθμίσεις για τη μετανάστευση προς την Τουρκία. Εδώ πάλι τα κράτη-μέλη πάνε να βρουν τα χρήματά τους στα προγράμματα τα καθοριστικά, αυτά τα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκής φύσεως. Και προσπαθούμε μεταξύ μας να τα βρούμε και να διατητεύσουμε κατά πόσο το Ταμείο για την Άμυνα, που είναι ένα Ταμείο Έρευνα και Ανάπτυξη, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στα πλαίσια του FP9. Γιατί, διότι δεν υπάρχουν πόροι. Γι' αυτό κάθομαστε και το συζητάμε. Ενώ κανεί ε, δεν συζητάει, ή πολύ λίγοι συζητάνε, εν περιπτώσει, ε, για το κατά πόσο αυτά τα προγράμματα είναι σκόπιμα ή όχι. Είμαστε λοιπόν πραγματικά στην καρδιά του προβλήματο εδώ. Η δυνατότητα του προπολογισμού να, προ, να προσπιστεί τι ε, προτεραιότητε ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί όπου η Ευρώπη μπορεί να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνουν τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί λοιπόν οι αποφάση που παίρνονται σε επίπεδο προπολογισμού ε, ε να είναι υπέρ ή κατά τη Ευρώπη, αλλά να είναι θέμα του κατά πόσο είμαστε υπέρ ή κατά του μέλλοντος της Ευρώπης. Ε, δεν μπορούμε ε, κοντόφθαλμα να βλέπουμε το μέλλον. Ε, η ανάπτυξη, η έρευνα, οι επενδύσεις, οι υποδομές, ε, ε, αυτά είναι τα ε, στοιχεία τα οποία περισπίζεται η Επιτροπή μας και αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Νομίζω ότι ουσιαστικά συμφωνώ και με αυτό που πάνε προαλήσαντες, Πρόεδρε. Είμαστε στο ίδιο, κινούμε στο ίδιο πνεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλουν και άλλοι συνάδελφοι το λόγο. Ο κύριος Ρούμπικ είναι στον κατάλογο ομιλητών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους συναδέρφους αποφασιστική σημασία στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο είναι να επικεντρωθούμε στον προϋπολογισμό και ιδιαίτερα στο πρόγραμμα Horizon 2020. Τον Δεκέμβριο αποδείξαμε ότι αν κάτσουμε μέχρι τις 4 το πρωί μπορούμε να βρούμε 100 ε, εκατομμύρια για το ε, ε, ορίζον 2020. Πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα πόσα όσα είναι διατεθειμένοι να δώσει το Συμβούλιο. Ενημερώθηκα ότι δεν θέλουν να συζητήσουν ε, ε, για οτιδήποτε πάνω από τα 100 εκατομμύρια, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε ζητώντας 250 εκατομμύρια λαμβάνοντας υπόψη το ε, συνολικό πρόγραμμα, δεν είναι και πάρα πολλά αυτά τα χρήματα. Και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το πρόγραμμα COSME και να βρούμε ε, δραστηριότητες ε, που να, να βρούμε δράσεις για την αγορά εργασίας. Τρίτη παρατήρηση. Αναφέρθηκαν ήδη οι οργανισμοί. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τι συνέργειες θα είναι δυνατές στο μέλλον. Να ενισχύσουμε την συνεργασία μεταξύ των ε, οργανισμών, για παράδειγμα του ΕΣΑ, της ΕΝΙΖΑ, του ΜΠΕΡΕΚ κλπ. Θα μπορούσαμε έτσι τουλάχιστον την τεχνική διεκπαιρέωση να τη διαμορφώσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Του χρόνου έχουμε ευρωεκλογέ. Το Ευρωπαρόμετρο μας δείχνει ότι οι άνθρωποι της Ευρώπης ε, βλέπουν ε, πιο χρήσιμα να είναι τα προγράμματα ε, έρευνας και επιστήμης. Εάν λοιπόν ε, είμαστε διατεθειμένοι να ε, παλέψουμε με το Συμβούλιο, αυτό είναι το πιο σημαντικό μας επιχείρημα, ότι έχουμε με το μέρος μας τους πολίτες. Πιστεύω λοιπόν ότι σκληρή γραμμή από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι ε, ο καλύτερος τρόπος να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ακούει κανείς τους συναδέλφους από την Επιτροπή Προϋπολογισμού, πραγματικά ανησυχεί. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πραγματικά εδώ έχουμε μια φυγή προς τα μπρος από το Συμβούλιο. Είναι πραγματικά ανεύθυνα τα κράτη-μέλη. Είμαι λίγο αυστηρή, αλλά έτσι είναι. Ζητάει όλο και πιο πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη, αλλά δεν θέλουν να ε, πληρώσουν γι' αυτό το ταμείο για το οποίο είμαι εγώ η συγκήτρια, το, ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για το 2019-2020. Είναι αποφασισμένο αυτό το ποσό, όλοι έχουμε συμφωνήσει γύρω από αυτό, αλλά δεν τα έχουμε βρει μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Και πραγματικά απογοητεύτηκα όταν χθε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, άκουσα τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κατάινεν, ε, της Κομισιόν να ζητάει από το Κοινοβούλιο να κάνει μια προσπάθεια στη διαπραγμάτευση του προπολογισμού. Και του απάντησα την προσπάθεια, η προσπάθεια πρέπει να γίνει από δύο πλευρές. Από την πλευρά του Συμβουλίου και από την πλευρά του Κοινοβουλίου, αλλά αυτό που πραγματικά είναι αδιανόητο είναι συστηματικά να πηγαίνουμε να παίρνουμε χρήματα από δημοσιονομικές γραμμές που έχουν να κάνουν με την οριζόντα 2020 ή με από άλλα κονδύλια που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Ανευθυνότητα λοιπόν σε μια στιγμή όπου υπάρχει μια στροφή στην κοινωνία μας προς τις νέες τεχνολογίες. Εάν δεν κάνουμε τις προσπάθειες, τις απαραίτητες προσπάθειες τώρα, τότε η καθυστέρηση αυτή θα συσσωρευτεί και σε 15-20 χρόνια θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά η ανευθυνότητα αυτή των κρατών μελών θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά τότε. Θα πρέπει λοιπόν ε, να είμαστε εξαιρετικά ενωμένοι ε, σε αυτή την ε, συζήτηση. Βεβαίω, στην σημαία διαπραγμάτευση όλοι πρέπει να κάνουν υποχωρήσει, αλλά η συμπεριφορά του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή με την υποστήριξη μάλιστα τη Κομισιόν είναι πραγματικά απαράδεκτη. Και θα πρέπει εκεί εμεί να είμαστε εξαιρετικά σκληροί στη στάση που θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Γκροστέτ. Όπως βλέπετε κύριε Σιγητά, είμαστε απολύτως ενωμένοι εδώ στην Επιτροπή Ήτρε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Είναι σαφή τα πράγματα, άλλωστε, μετά από αυτά που ακούστηκαν εδώ στην Επιτροπή μας. Και τώρα θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια σχόλια και από σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πράγματι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, ε, τα σχόλια και ε, γιατί εντός του Κοινοβουλίου, ακόμη και αν εργαζόμαστε σε διάφορες επιτροπές, είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι. Εγώ είμαι ικανοποιημένο που θα ήθελα η δική σας επιτροπή να εκπροσωπείτε καλά Μάλλον χαίρομαι που η Επιτροπή σε εκπροσωπείται τόσο καλά από τον κύριο Γκάιερ ε, στην Επιτροπή Προπολογισμού όπως και από τον συνάδελφο Ρούμπιχ με τον οποίο κάνουμε μαζί τη συνδιαλλαγή εδώ και χρόνια χωρίς ε, να μπω στην ουσία απλώ θα σχολιάσω το πολιτικό σκέλος ότι ε, είπα, πρέπει ε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, Επιτροπής. Ε, ακούσαμε τον κύριο Κατάνιν που ζήτησε να κάνει μια προσπάθεια το Κοινοβούλιο, όμως ε, πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιό να πει στο Συμβούλιο να κάνει αυτό μια προσπάθεια. Και το Συμβούλιο πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε εμά γιατί εκπροσωπούμε την κοινωνία των πολιτών. Αλλά πάντοτε εμείς ε, ουσιαστικά απαντάμε σε πραγματικά αιτήματα που προέρχονται από τους πολίτες. Αυτά που ζητούμε εμείς δεν τα ζητάμε για την δική μας επιθυμία, αλλά προκύπτει από την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πολίτες. Εμείς πρέπει να ε, έχουμε αυτή την αρχή η οποία θα μας καθοδηγεί. Θα είμαστε ενωμένοι λοιπόν ε, επ' αυτής της αρχής και ε, πρέπει να υποστηρίξουμε ότι θέλουμε νέα προγράμματα με νέε χρηματοδοτήσει. Δεν μπορούμε να έχουμε νέα προγράμματα χωρί νέα χρηματοδότηση, γιατί όπω είπατε είναι σφιχτό ο προπολογισμό. Ήδη όλα έχουν ε, κατανεμηθεί και για το επόμενο έτος, αλλά και για τα επόμενα έτη, για τα μελλοντικά έτη. Κάτι τελευταίο ε, που θέλω να ζητήσω ως πολιτικός ε, παρά ως ε, γενικός εισηγητής προϋπολογισμού. Αυτό που θέλω να ζητήσω είναι ο καθένας από εμά ε, να κάνει μια προσπάθεια στη χώρα του με τη δική του κυβέρνηση. Γιατί κατόπιν βρισκόμαστε ενώπιον του Συμβουλίου που ε, ουσιαστικά όπου ουσιαστικά εκπροσωπούνται κυβερνήσει, όμω θα πρέπει οι δικέ μα εθνικέ κυβερνήσει να είναι πεπισμένε για αυτά που λέμε. ίσως ε, ε, θα έπρεπε και εμείς να διαδραματίσουμε ένα τέτοιο ρόλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και μια πιο ήπια θέση από την πλευρά του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής. Σας ευχαριστούμε για τις ε, παρατηρήσεις σας, τις καταληκτικές. Είναι πολύ σημαντικό να αισθανόμαστε ότι έχουμε Φίλου στην ομάδα προπολογισμού και ότι έχουμε κοινέ προτεραιότητε. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ενώπιον μα μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Σήμερα Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για την επιστολή στην Επιτροπή Προπολογισμού σε σχέση με τις προτεραιότητε της ΣΥΤΡΑ για τον προπολογισμό του 2019. Και στις αρχές Ιουνίου 2018 θα αποστείλουμε αυτή την επιστολή, περίπου σε ένα μήνα και κάτι. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα ως μέλη της Επιτροπής ΙΤΡΕ να προτείνουμε τροπολογίες για τις γραμμές του προπολογισμού. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στην Επιτροπή Προπολογισμού είναι 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου λοιπόν και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 10 Ιουλίου στην Επιτροπή Προπολογισμού. Συγγνώμη, στην Ήτρε, διορθώνει ο Πρόεδρος, στην Ήτρε. 10 Ιουλίου θα έχουμε την ψηφοφορία. Τρίτη διαδικασία. Γνωμοδότηση της Ήτρε για το ψήφισμα για τον προπολογισμό του 2019 και εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης θα γίνει στις 10 Ιουλίου στην Επιτροπή Ήτρε, 10 Ιουλίου. Επομένως έχουμε την ίδια ημερομηνία με την ψηφοφορία στην Ήτρε για τις τροπολογίες για τις γραμμές του προπολογισμού. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για την γνωμοδότηση 5 Σεπτεμβρίου και ψηφοφορία της Ήτρε επί της γνωμοδότησης 24 Σεπτεμβρίου. Έχουμε λοιπόν τρεις παράλληλες διαδικασίες. Την επιστολή αρχές Ιουνίου θα τη στείλουμε. Τροπολογίες για τις γραμμές του προπολογισμού. Θυμηθείτε ότι τον Ιούνιο θα πρέπει να τις καταθέσουμε και θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο και η γνωμοδότηση της Ήτρε θα την ψηφίσουμε στις 24 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους από την Επιτροπή Προπολογισμού που ήταν εδώ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο αυτό και πάμε στο σημείο 13. Ε, πρόγραμμα έρευνα και εκπαίδευση τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντα 2020. Η συγγήτρια είναι η Ρεμπέκα Χάρμ. Ε, έχουμε και ένα σχέδιο έκθεση εδώ μπροστά μα. Ε, το πρόγραμμα κατάρτισης της Euratom ε, για την έρευνα από το 2014 ε, θέλουμε, η πρόταση είναι να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα το 2019 να υπάρχει μια συνέπεια των δράσεων καθ' όλης διάρκειας του επταετούς προγράμματος. Ε, αγαπητή Ρεμπέκα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Γέζρι. Θα μιλήσω γερμανικά, είναι πιο εύκολα για μένα, ειδικά για αυτό το θέμα. Ως εισηγήτρια, όπως μπορείτε να δείτε και στο σχέδιο έκθεσής μου, Είμαι της άποψης ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά καθήκοντα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης και θέλω να ε, αλλάξουμε επίκεντρο στο μέλλον ε, στο πρόγραμμα αυτό. Πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να ασχοληθούμε με, με την ε, πρόκληση των ε, παλαιών πυρηνικών εργοστασίων ε, καθώς ε, και με το θέμα της ε, διαχείρισης των αποβλήτων. Αυτό το έχω καταστήσει σαφές στην έκθεσή μου. Και επίσης όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα αυτό μας περιμένουν σημαντικές προκλήσεις. Αυτά προκύπτουν και από τις συζητήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω στο θέμα αυτό. Φαίνεται λοιπόν σαφώς ότι έχουμε ανάγκη από ε, ε, εξειδικευμένο προσωπικό ακόμα και στις χώρες ε, που έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει το σημαντικό θέμα της ε, αποθήκευσης των αποβλήτων. Κάποια κράτη-μέλη χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια εδώ και 50 χρόνια και παρόλα αυτά όσον αφορά την τελική διάθεση των αποβλήτων δεν έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα. Η Γερμανία πριν μερικά χρόνια αποφάσισε να ξεκινήσει από την αρχή την αναζήτηση κατάλληλου χώρου τελικής αποθήκευσης. Ε, στην Σουηδία υπάρχει ένα αρκετά ε, προχωρημένο πρόγραμμα, το οποίο όμως σταμάτησε ε, με δικαστική απόφαση που ζητάει επανεξέταση όλων των τεχνικών στοιχείων. Δεν καταφέρνουμε λοιπόν να βρούμε μέρη τελικής αποθήκευσης των αποβλήτων αυτών, ενώ υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το πρόβλημα αυτό. Αυτό που συνδέει τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους είναι ότι δεν έχουν επαρκή χρηματοδότηση για τον ε, παροπλισμό των πυρηνικών εργοστασίων ε, και για την ε, τελική αποθήκευση των αποβλήτων. Θα πρέπει λοιπόν ε, στον τομέα της έρευνας ε, να δώσουμε βάρος ε, στα θέματα αυτά. Όσον αφορά τον διαχωρισμό και τη μεταστοιχίωση, και εδώ δεν βλέπω να υπάρχουν σημαντικές πρόοδοι. σε άλλους ε, τομείς ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα εάν συγκεντρώσουμε πόρους για την έρευνα. Το πρόγραμμα της Ευρατόμ ε, δεν θα πρέπει να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες αντιδραστήρων και και για την διάσπαση του ατόμου αλλά και για την σύνδεξη ισχύουν τα ίδια. Έχουμε μιλήσει για τη χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ, το οποίο όμως εδώ δεν αμφισβητείται. Ε, είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά. Με οποιονδήποτε και να μιλήσει κανείς για το ΙΤΕΡ και για την τεχνολογία σύνδεξης, ε, ένα είναι απόλυτα σαφές. Αυτή η πολύ δαπανηρή έρευνα δεν θα συμβάλλει ε, στην επίλυση των ε, προβλημάτων μας όσον αφορά το κλίμα, διότι η εμπορική χρήση της ε, σύνδεξης προβλέπεται για πολύ μετά το 2050 έτος κατά το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσουμε αποτελέσματα όσον αφορά το κλίμα μας. Ε, οι εμπειρογνώμονες ε, σήμερα δεν ε, βάζουν ημερομηνία στην εμπορική χρήση της σύνδεξης. Στις έρευνες πάνω στην διάσπαση του ατόμου, Πιστεύω ότι τα ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει να διαμορφωθούν με δίκαιο τρόπο για όλα τα κράτη-μέλη. Περισσότερα από τα μισά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ πυρηνική ενέργεια είτε έχουν ε, λάβει αποφάσεις εγκατάλειψής της. Και γι' αυτό η δική μου πρόταση είναι να μεταφέρουμε αλλού το κέντρο βάρους του ερευνητικού αυτού προγράμματος, να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα και να εξετάσουμε πτυχές ασφαλείας και διάθεσης πυρηνικών αποβλήτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για το σχέδιο έκθεσή σας και τις απόψεις που μας παρουσιάσατε. Σκιώδης εισηγητές. ΕΛΚ, ο κύριος Ουρούτσεφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Χάρμς, η οποία στην έκθεσή της ε, σαφώς περιγράφει ε, τις, το που βρίσκονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πυρηνική ερεύνα, ιδιαίτερα τα ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας και τα διάφορα project ε, σχετικά με την πυρηνική σχάση. περίπου η μισή καθαρή ενέργεια, δηλαδή χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, είναι πυρηνικής προέλευσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πυρηνικά εργοστάσια ε, υπάρχουν, λειτουργούν εδώ και δεκαετίες ε, και είτε δημιουργούμε νέα πυρηνικά εργοστάσια είτε παρατείνουμε το χρόνο ζωής των προηγούμενων. Είναι λοιπόν αναγκαίο να συνεχιστεί η έρευνα για την υποστήριξη της ασφαλούς εκμετάλλευσης της πυρηνικής ενέργειας στα ίδια επίπεδα με τα τωρινά. Ιδάλω δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα ασφάλεια με βάση και την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια. Η προτινόμενη λοιπόν ε, μείωση ε, της πυρηνικής ε, έρευνας είναι απαράδεκτη αυτή τη στιγμή. Αυτές τα δραστηριότητες στα πλαίσια της Euratom και του σχετικού ερευνητικού προγράμματος προχωρούν κυρίως στα πλαίσια διεθνών συνθήκων και πρωτοβουλειών όπου συμπετέχουν οι πιο προηγμένες τεχνολογικά χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι Καναδά, ο Καναδάς πρόσφατα εξέφρασε ενδιαφέρον για να συμμετάσχει στο σχέδιο ITER διότι η περίπλοκη έρευνα που έχει να κάνει με την πυρηνική ε, σχάση ως ε, πηγή ενέργειας ε, απαλλαγμένη από άνθρακα συνοδεύεται από μια σειρά τεχνολογικές ε, εφευρέσεις, ανακαλύψεις, ε, διαδικασίες. Ε, είναι δύσκολο να κάνουμε τώρα μια αξιολόγηση ή να εξετάσουμε την εμπορική πτυχή του ζητήματος. Ούτε μπορεί το πρόγραμμα έρευνας της Euratom για το 19-20 να μπορέσει να συμπεριλάβει διεθνή project στα πλαίσια της πυρηνικής χάσης όπου είναι σε ηγετική θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχιστεί η πυρηνική έρευνα για τα επόμενα δύο έτη είναι λογική. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες που υπάρχουν ε, σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια και ανταποκρίνεται και στις διεθνείς δεσμές που έχουμε αναλάβει. Πρέπει λοιπόν να τύχει υποστήριξη χωρί σημαντικέ τροπολογίε ή ε, Μάλιστα. Εκ μέρου των Σοσιαλιστικών και και Δημοκρατών, ο κύριος τη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για το έγγραφο. Εγώ σέβομαι την άποψή σα αντιλαμβάνομαι ότι είστε κατά τη πυρηνική ενέργεια, όμω ε, ω εκ ως εισηγητής για το S&D πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ μαζί σας. Το σχέδιο κανονισμού αναφέρεται στην επέκταση ενός ήδη υπάρχοντος προγράμματος έρευνας και ε, καινοτομίας ε, ε, για δύο χρόνια ακόμα και αυτό είναι λογικό ε, διότι πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν είναι ένα καινούριο πρόγραμμα. Πρέπει να ολοκληρωθεί το προηγούμενο πρόγραμμα. Και όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια, θέλουμε να βρούμε ε, ασφαλείς αναλλακτικές σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση των αποβλήτων και θέλουμε να αναπτύξουμε και ε, πυρηνική τεχνολογία στο φαρμακευτικό τομέα. Επίσης υπάρχει το θέμα της σχάσης. Πιστεύουμε ότι το μέλλον τεχνολογία θα μας επιτρέψει ε, να παράγουμε επαρκή ενέργεια και η πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη. Στη χώρα μου, παραδείγματος χάρη, αγοράζουμε ε, ενέργεια, εισάγουμε ενέργεια από άλλες χώρες. Και συνήθως αυτή η ενέργεια παράγεται σε πυρηνικά εργοστάσια. Ξέρουμε ότι είναι η πιο φτηνή και η πιο καθαρή ε, μορφή ενέργειας. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ασφάλεια ε, και χρειαζόμαστε μεγαλύτερο συντονισμό και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, θα γίνει με ασφαλή τρόπο ε, η, ε, η απόσυρση κάποιων εργοστασίων έχουμε ένα παλιό σοβιετικό αντιδραστήρα εμείς ε, και παίρνει χρόνο η διαδικασία ε, κλεισίματος του, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται συντονισμός, πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Είναι σημαντικά και χρήσιμα αυτά τα βήματα για τις χώρες που προσπαθούν ε, να κλείσουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Θα πρέπει ε, να προωθήσουμε την ασφαλή διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, αλλά ε, δεν συμφωνώ μαζί σας που ε, ε, ζητάτε να διαγραφεί από την πρόταση, να διαγραφούν μια σειρά από σημαντικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, αυτή την τεχνολογική, την τεχνική σχάσης. Το σχέδιο αυτό είναι σημαντικό την τεχνική σύνδεξη με συγχωρητό και σχάσεις. Πιστεύω ότι μόνο η έρευνα θα μπορέσει να εξασφαλίσει ότι η ενέργεια σύνδεξης θα ε, αποτελέσει ε, μια ασφαλής πηγή ενέργειας στο μέλλον. Θα μας βοηθήσει αυτό να, να καλύψουμε τις ανάγκες μας ε, σε ένα περιβάλλον ενεργειακής ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε και τη νέα παραγωγή Καθαρή και ασφαλού ενέργειας στο μέλλον. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στι ανανεώσιμε πηγέ. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η θέση μας στην παγκόσμια αγορά για να μείνουμε ανταγωνιστικοί. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αυτό το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης. Ε, ε, η ομάδα μου λοιπόν θα υποστηρίξει το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ των Φιλελευθέρων, κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την συγγήτρια για το έργο της. Όταν μιλάμε για ατομική ενέργεια, για πυρηνική ενέργεια, ουσιαστικά μιλάμε για κάτι ιερό. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν απολύτως την πυρηνική ενέργεια, ενώ ε, κάποιοι άλλοι έχουν λάβει κάποιες ριζοσπαστικέ θέσει απέναντι στο θέμα. Όταν είμαστε κατά της πυρηνική ενέργειας ε, θέλουμε να τη θάψουμε και όχι μόνο να θάψουμε τα τελικά απόβλητα αλλά ολόκληρο τον τομέα. Και υπάρχουν βέβαια και άλλοι που πιστεύουν ότι πρέπει να την υποστηρίξουν. Έχουμε λοιπόν αντιδιαμετρικά αντίθετες θέσει. Ε, τώρα, η εισηγήτρια έχει, καθώς ε, δεν υποστηρίζει τη συνέχιση της πυρηνικής ενέργειας, ε, έχει ε, οδηγεί στην έκθεση προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως στον τομέα και στη διάρκεια ζωής της πυρηνικής ενέργειας φτάνουμε να την ξεφορτωθούμε και έτσι να επιλύσουμε μία σειρά προβλημάτων. Εξού και το θέμα της πιστότητας στο πρόγραμμα που είναι ένα πιο ευρύ πρόγραμμα. Έχει ως στόχο να βελτιώσει την ανάπτυξη, να ε, προωθήσει την ασφαλή έρευνα και τα λοιπά. Οι άλλες ομάδες ε, υποστηρίζουν ε, την πρόταση της Κομισιόν και είμαστε εδώ στην εξής ε, κατάσταση. Ε, δηλαδή, εμείς ε, σκοπεύουμε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα και να υπάρχει χρηματοδότηση μέχρι το 2019. Κάποιες παρατηρήσεις όμως έχω παρόλα αυτά. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρηνικής ενέργειας, απέναντι στην ανθρώπινη υγεία. Να επισημάνω ότι η πυρηνική ενέργεια έχει προκαλέσει πολύ λίγα θύματα σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας. Ξέρετε πολύ καλά ότι και εγώ προέρχομαι από μια χώρα με εξορρυκτική διαδικασία, με ορυχία και είχαμε ε, στην διαδικασία της εξόρυξης ε, χιλιάδες ε, νεκρούς. Δεν μιλάω τώρα για τις εκπομπές και για το κλίμα. Και η πυρηνική ενέργεια ήταν η πιο ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία. Όμως ο πιθανός κίνδυνος μας φαίνεται πολύ μεγάλος ως προς την κλίμακα, γι' αυτό ουσιαστικά γίνεται σχεδόν κάτι ιερό το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. ό,τι αφορά την ε, κατάρτιση και την έρευνα. Ε, μπορούμε να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και πώς επηρέαζεται την ανθρώπινη υγεία. Δεν ε, νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέλλον, όμως νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ πιο σημαντικό. Εγώ πιστεύω στη σύνδεξη και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί Πιστεύω ότι θα κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε και αν δούμε τα μεγάλα προγράμματα έρευνας, ίσχυε κάτι τέτοιο για την σχάση, ισχύει και για τη σύνδεξη. Και πιστεύω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις μέχρι το 2050. Σήμερα ε, αλλού στον κόσμο η πυρηνική ενέργεια μέσω της σχάσης ε, είναι κάτι που χρησιμοποιείται. Έχουμε πάνω από 240 αντιδραστήρες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή παγκοσμίω. Και ενώ εμείς είμαστε ε, σημαντικοί παίκτες, θα αποφασίσουμε ότι θα μείνουμε εκτός αυτής της διαδικασίας. Δεν μου φαίνεται να είναι και πολύ ρεαλιστικό. Επομένως, εμείς είμαστε κοντά στη θέση της Κομισιόν. Θέλουμε να συνεχιστεί η υποστήριξη στο πρόγραμμα αυτό. Και μια τελευταία λεπτομέρεια σε σχέση με το θέμα της ισότητας ε, των δύο φύλων ε, στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης. Ε, είναι ένα θέμα απέναντι στο οποίο έχω θετική στάση. Γιατί ξέρετε η κατάρτιση των επιστημόνων ε, εμφάνιζε κάποιες ανισότητες στο παρελθόν, επομένως υποστηρίζω αυτή την πτυχή. Βέβαια, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το προσωπικό στα προγράμματα έρευνας και κατάρτισης. Τώρα βέβαια το αν ε, θα εγκαταλείψουμε την πυρηνική έρευνα για να περάσουμε στην κβαντική, αυτό είναι ένα ζήτημα που μου φαίνεται μη ρεαλιστικό. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Ηλικιώτης θα αντικαταστήσει την κυρία Ματίας, που δεν είναι εδώ. Από την ΚΟΕ βέβαια και οι δύο. Έχετε το λόγο κύριε Σιλκιώτη. Πρόεδρε, ε, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Ρεβέκα Χάρμς για την έκθεση που έχει καταθέσει. Όπως είπατε, η σκιώδη συζητήτρια μας δυστυχώς δεν βρίσκεται στις Βρυξέλλες, γι' αυτό που ζήτησε να την αντικαταστήσω. Για την QNGL είναι ξεκάθαρο πως η πυρηνική ενέργεια ενέχει τεράστιους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται για ειρηνικούς σκοπούς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενισχυθεί περισσότερο η έρευνα για ενίσχυση της ασφάλειας που αφορά την πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, το νομίζω πω συμμεριζόμαστε την άποψη πω δεν πρέπει να χρηματοδοτείται η πρόθεση τη έρευνα για συντήρηση των μονάδων πυρηνική ενέργεια. Οι προτεραιότητε μα πρέπει να είναι να προωθούν νέε μορφέ ενέργεια, η καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια. Προ την ίδια κατεύθυνση θεωρούμε πω πρέπει να πάψει η στήριξη που δίνεται σε οργανισμού όπω ο ΙΤΕΡ, που προωθεί την πυρηνική ενέργεια και ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να απογραμμίσω πω για την ομάδα μα είναι σημαντικό να προωθείται και να χρηματοδοτείται η έρευνα και η κοινοτομία που στόχο έχει την εξυπηρέτηση των συμφωνών και των αγκών τη κοινωνία, του ανθρώπου και το περιβάλλον. Ευχαριστώ, πολύ. Uh, thank you, colleague, for your remarks and uh, uh, presentation. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Εκ μέρους κυρία Λεσσεβαλιέ. Θα την καταστήσει την κυρία Κάπελ ως και οδησηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην πρώτη μου παρέμβαση είχα υπογραμμίσει ότι υποστηρίζω το όραμα της Κομίσιον που θεωρεί την πυρηνική ενέργεια ως χρήσιμη πυρηνική ενέργεια για τη μείωση των εκπομπών. Είχα δηλώσει ότι ήμουν ικανοποιημένη με το κείμενο που είχε προτείνει η Κομισιόν και ως ε, και η συγγήτρια να προσπαθήσει να βρει μια ενδιάμεση θέση. Όμως διαπιστώνω ότι δεν προσπαθήσατε να βρείτε ε, ουσιαστικά ένα πεδίο συνεννόησης μεταξύ των διάφορων ομάδων και μεταξύ των εθνών που έχουν κάνει διαφορετικές επιλογές ε, για το για την πυρηνική ενέργεια. Παρουσιάζετε τις θέσεις της ομάδας σας ε, κατά της πυρηνικής ενέργειας και τις επιλογές της χώρας σας. Έτσι λοιπόν φαίνεται ε, να ε, θεωρείται την ε, Ευρατό ως έναν οργανισμό διάλυσης, παροπλισμού της πυρηνικής ενέργειας. Εμείς τώρα να σας πω ότι κατασκευάζουμε και ένα νέο αντιδραστήρα Θέλουμε ο, οργανισμός να θέσει ως προτεραιότητα την διάθεση των πυρηνικών απευλήτων, όμως δεν θα πρέπει να πληγεί η έρευνα και η κατάρτιση θεωρείται ότι είναι ξεπερασμένη η πυρηνική ενέργεια, όμως δεν ισχύει κάτι τέτοια και η έρευνα ε, σε αυτή ε, την μορφή ενέργειας θα πρέπει να συνεχιστεί, καθώς έχει χαμηλές εκπομπές. Επίσης, ε, Εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει η ευρωτόμη να συνεχίσει να διατηρεί τις εργασίες έρευνας. Εμείς ε, ανανεώνουμε την υποστήριξή μας στην έρευνα για την ενέργεια σύνδεξης. Εσείς στο κείμενό σας θέλετε να διαγράψετε κάθε αναφορά. Αυτό το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα είναι παράδειγμα συνεργασίας που ενώνει τα ευρωπαϊκά έθνη και τις ε, κύριες παγκοσμίες δυνάμεις που αποτελούν πάνω από το ίμιση της ανθρωπότητας. Επιπρόσθετα. Ε, μόνιμες χρηματοδοτήσεις ε, στο μέλλον ε, θα πρέπει να δοθούν το να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο όραμα νομίζω ότι είναι απαραίτητο σήμερα και κάτι τελευταίο για να υποστηρίξουμε την αναφορά που κάνετε στην τρομοκρατική επιλή το να, να κατασταθούν ασφαλή τα πυρηνικά εργοστάσια απέναντι σε αυτή την απειλή είναι κάτι πολύ σημαντικό και ελπίζουμε να μην αποτελεί μια απλή φράση στο κείμενό σας. Σας ευχαριστούμε για τις ε, παρατηρήσεις σας εκ μέρους του ΙΕΝΕΦ. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγοντα του συναδέλφου, ε, πιστεύω ότι η δουλειά τη ισχύτριας θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη, διότι και εγώ θεωρώ ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παράταση για δύο έτη του προγράμματο πλαισίου έρευνα τη Euratom είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Θέλω να θυμίσω, το είπαν και άλλοι συναδελφοί, ε, ότι η πυρηνική ενέργεια είναι κεφαλαίου σημασίας, ε, μιας και δεν περιέχει άνθρακα. Ε, δεν πρέπει λοιπόν εδώ να αρνούμαστε την πραγματικότητα και να λέμε ότι δεν χρειαζόμαστε την, την πυρηνική ενέργεια στον τομέα της ε, υγείας. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την έρευνα την ευρωπαϊκή στον, στον πυρηνικό τομέα και να υπάρχει μια συνέχεια. Πρέπει να είμαστε συνεπείς ε, στην ατζέντα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αντίθετα με την εισηγητρία, θεωρώ ότι να μειωθεί ο προπολογισμό για αυτό το πρόγραμμα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αποτελεί μέρο των κονδυλίων που προβλέπονται για την περίοδο 2014-2020. Τώρα βέβαια όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε ε, ε, να προσπαθήσουμε ε, να έχουμε μια ασφαλή αποπυρηνικοποίηση των παρόν εργοστασίων Υπάρχει όμως και το θέμα τεχνολογικής ε, ηγεσία, ε, να είμαστε στην πρώτη γραμμή δηλαδή. Μιλήσαμε για το ΙΤΕΡ, για, τους, για νέα συστήματα αντιδραστήρων, το σύνολο του κύκλου ε, των, του, των πυρηνικών καυσίμων. Βεβαίως κάποιοι επιστήμονε θεωρούν ότι δεν θα υπάρχει στο μέλλον εμπορική εφαρμογή σε 50 χρόνια της πυρηνικής σύνταξης. Αν δούμε τι λέγανε οι επιστήμονες πριν από 50 χρόνια, ε, κανείς δεν είχε προβλέψει αυτά που θα συνέβαιναν. Ε, η ε, τεχνητή νοημοσύνη και μια σειρά από νέες τεχνολογίες που συζητούμε εδώ στην Επιτροπή μας. Θα σταματήσουμε λοιπόν ε, να ακούμε επιστήμονες που σε 50 χρόνια που δεν θα είμαστε εδώ εμείς βέβαια δυστυχώς αλλά θα πρέπει να προετοιμάσουμε για, το, για τους νέους το μέλλον και είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την έρευνα στα πλαίσια του Ευρατόμ. Ευχαριστώ. Uh, uh, thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μούντι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Είναι μια από τις σπάνιες περιστάσεις που βρίσκομαι να διαφωνώ με την εισηγήτρια και συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες, σχεδόν όλους τους προλαλήσαντες. Όσον αφορά το πού βρίσκεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη γενική υποστήριξη αυτής της θέσης. Φυσικά η διαχείριση των αποβλήτων και ο παροπλισμός είναι πολύ σημαντικά θέματα, αλλά αυτά αποτελούν ήδη μέρος της πρότασης που συζητάμε. Και υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία στο κείμενο ε, πάνω στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά νομίζω σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που προτείνει η συγγήτρια. Για παράδειγμα, την εκπαίδευση και κατάρτιση ε, για τις ε, πηγές ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, την εκπαίδευση και την έρευνα, την κινητικότητα. Όσον αφορά το ίτερ, πρόκειται για ένα διεθνές ε, πρόγραμμα και πρέπει να είμαστε περήφανοι που ηγούμαστε σε αυτό και που ήδη παρέχει νέες τεχνολογίες ε, και τεχνολογικές εξελίξεις και όσον αφορά ε, τα υλικά και τεχνολογίες χειρισμού εξ αποστάσεως. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να διευθύνουμε αυτό το πρόγραμμα. Και κάποιες ακόμη παρατηρήσεις. Καταρχάς, να φροντίσουμε να συνεχίσουμε την ε, δουλειά μας ε, πάνω στο θέμα αυτό, μεταξύ άλλων ε, και το κοινό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και το άλλο θέμα είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την συνέχιση του προγράμματος αυτού. Τέλος, ε, θα διαφωνήσω με τον συνάδελφο τη Άλτε όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει πάντα να είναι... Ε, να, να διέπει τις εργασίες μας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε οι γυναίκες να έχουν όσο περισσότερες θέσεις σε τέτοια προγράμματα. Πάντως ε, νομίζω και εγώ ότι θα πρέπει να επιλέξουμε άλλη κατεύθυνση από αυτή που προτείνει η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χένκελ μήπως θέλει κάτι να προσθέσει. Διότι είστε σκιώδης εισηγητής. Ναι, ζητώ συγγνώμη, δεν μπόρεσα να είμαι παρόν, διότι είχα υπουργό εξωτερικών στο γραφείο μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εισηγήτρια της Ήτρε, η κυρία Χάρμς, επιλέγει άλλη κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιλάει πάντα για παροπλισμό των πυρηνικών εργοστασίων στην έκθεσή της. Αυτό το βλέπω σε πολλές από τις προτινόμενες τροπολογίες. Σε πολλές περιπτώσεις προτείνει τη διαγραφή φράσεων που τονίζουν το ρόλο της πυρηνικής ενέργειας και της σχετικής έρευνας στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίζουν τι είδους ενέργεια θέλουν να ε, χρησιμοποιούν και όχι να προσπαθούμε να επιβάλλουμε τη γερμανική λύση, για παράδειγμα, σε χώρες σε κυρίαρχες. Και όταν μιλώ για τις γερμανικές λύσεις ε, πρέπει μάλλον να αναφέρομαι σε ε, λύσεις των ε, γερμανόφωνων χωρών, Αυστρίας και Γερμανίας. Καμία χώρα δεν θέλει να ε, εξαρτάται απολύτως από την πυρηνική ενέργεια. Είναι σημαντικό όμως να βρούμε το σωστό ενεργειακό μείγμα για να έχουμε το πιο αποτελεσματικό προ προς το κόστος και το όφελος αποτέλεσμα μείωση της χρηματοδότησης ε, θα ε, είναι εις βάρος της ε, ηγετικής θέσης παγκοσμίως που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις πυρηνικές ενέργειες και θα εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να δημιουργεί εργαλεία για ασφαλή και καθαρή πυρηνική ενέργεια. Εάν θέλουμε να είμαστε η οικονομική και τεχνολογική δύναμη, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε όλους τους τομείς έρευνας και τεχνολογίας και θα πρέπει να μπορούμε να διαφοροποιούμαστε και να ανταγωνιζόμαστε σε όλους τους τομείς. Εάν όχι, τότε η Ρωσία ή η Κίνα θα συμπληρώσουν το κενό αυτό που θα δημιουργήσουμε. Αυτό θέλουμε. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ηνωμένο Βασίλειο πάνω στην έρευνα μετά το Brexit. Έχω πει επανειλημμένα σε τούτη την αίθουσα, σε αυτή την Επιτροπή, αλλά και γενικότερα στο Κοινοβούλιο, ότι το Brexit είναι ένα τεράστιο λάθος. Ε, μόνο χαμένοι θα βγουν, θα βγουν από αυτήν την υπόθεση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα χάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να σημειώσουμε το γεγονός ότι φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διατεθειμένο να πληρώσει για τη συνέχιση της συνεργασίας μας στην έρευνα. Είχα συνάντηση με εκπροσώπους 15 Βρετανικών πανεπιστημίων και όλοι φαίνεται να συμφωνούν μαζί μου ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να συνεχιστούν όλα τα ερευνητικά προγράμματα που έχουμε και μετά το Brexit και ανησυχώ διότι οι προτάσεις ε, που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν αντικατοπτρίζουν αυτήν τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να υποβάλω τροπολογίες ε, για να τονίσω αυτό το θέμα που πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφα για τις παρατηρήσεις σας. να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Ζόλιφ Ποτρέλ, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την άποψη ε, που αναφέρεται στο σχέδιο έκθεσης ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα μπορεί να βελτιώσει την πυρηνική ασφάλεια ε, και την προστασία από την ακτινοβολία. Επίσης ε, σημειώνουμε ότι υπάρχει μια γενική υποστήριξη για την επέκταση του προγράμματος Ευρατόμ για την περίοδο 2019-2020. Αυτό εξέφρασαν τα μέλη που πήραν το λόγο στην προηγούμενη συνάντηση της Επιτροπής Ήτρε το Μάρτιο, όπως, αλλά και σήμερα όπως διαπιστώσαμε. Είναι προφανές ότι η συνένεση μετά τη Φουκουσίμα, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στα δύο στις προτεραιότητες των δύο προγραμμάτων για τα πυρηνικά μετά από το ατύχημα του 2011 εξακολουθεί να ισχύει. Το προτινόμενο πρόγραμμα για το 2019-2020 δίνει έμφαση στην πυρηνική ασφάλεια και των δικλειδών ασφαλείας με τους ίδιους βασικούς στόχους, τους ίδιους κανόνες. Γι' αυτό το λόγο, σε ό,τι αφορά την πυρηνική ασφάλεια και την έρευνα στον τομέα αυτών, θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ακριβώς τις ίδιες προτεραιότητες. Σε σχέση τώρα με τη σύνδεξη, η πρόταση υποστήριξης έχει να κάνει με μια στρατηγική που ε, αναφέρεται λεπτομερώς στον οδικό χάρτη για την πυρηνική σύνδεξη. Ε, θα πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν για διάφορους λόγους. Πρώτον για να προετοιμάσουμε την Ευρώπη για την εκμετάλλευση του ΙΤΕΡ. Δεύτερον για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια επιστροφή από την επένδυση αυτή σε αυτόν τον δύσκολο τομέα και για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιστήμης. Τρίτον, η Ευρώπη θα παραμείνει στο σωστό δρόμο για τη δημιουργία ε, των νέων πυρηνικών εργοστασίων. Δεν ξέρουμε αν η σύνδεξη τελικά θα παράγει ενέργεια για την ενεργειακά μας συστήματα. Είναι όμως ε, καθήκον μας προς τις μελλοντικές γενιές να εξετάσουμε επιστημονικά κατά πόσο αυτή η, η ενέργεια σύνδεξης είναι μια βιώσιμη πηγή ε, ηλεκτρισμού. Εάν ε, αποσυρθούμε τώρα, αυτό διακυβεύει το μέλλον και την προσπάθεια που γίνεται για μια ενέργεια χωρίς άνθρακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έχετε δύσκολο έργο, αγαπητή εισηγήτρια, όπως είπε και η κυρία Γκροστέτ προηγουμένως. Πώς τα βλέπετε εσείς. Εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις, λέει η κυρία Χάρμς. Όσον αφορά τον ΙΤΕΡ καταρχάς η πρώτη ε, έκθεση για την οποία ήμουν αρμόδια ως ε, βοηθός ε, στο Ευρωκοινοβούλιο τη δεκαετία του 80 είχε να κάνει με το ΙΤΕΡ και την δυνατότητα χρήση της πυρηνικής σύνδεξης μέχρι την αλλαγή του αιώνα, δηλαδή ανάμεσα στο 1995 και το 2000. Μερικοί συνάδελφοι θέλουν να πιστεύουν ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά την σύνδεξη σύντομα, αλλά αυτούς απλά μπορεί κανείς να ε, τους ε, χαϊδέψει ελαφρά στην πλάτη και να τους πει υπομονή, διότι από τότε που βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο συζητιέται η εμπορική χρήση της σύνδεξης από τους εμπειρογνώμονες. Ε, και αναβάλλεται συνεχώς η ημερομηνία, τώρα έχουμε φτάσει στα τέλη του παρόντος αιώνα. Υπάρχουν ε, άνθρωποι όμως που πιστεύουν βαθιά στην τεχνολογία αυτή. Αυτό που είναι βέβαια είναι ότι είναι οι ακριβότερες έρευνες στον τομέα της ενέργειας που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτόν και μόνο το λόγο λέω ότι πολύ χρήσιμη η βασική έρευνα, αλλά αυτά που γίνονται στο ίτερ πολύ γρήγορα ξέφυγαν από το πεδίο της βασικής έρευνας. οι περισσότεροι ευρωβουλευτές της Επιτροπής μας φαίνεται να μην έχουν ενημερωθεί από τους ίδιους τους επιστήμονες σχετικά με την εμπορική χρήση της ε, σύνδεξης. Ε, οι επιστήμονες ε, βρίσκονται υποπίεση από τον πολιτικό χώρο, αλλά δεν θέλουν να αναφέρουν συγκεκριμένη ημερομηνία για την εμπορική χρήση της σύνδεξης. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε πρότυπα ασφαλείας ε, που να ανταποκρίνονται στην, ε, στις τελευταίες ε, επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις. Όσον αφορά την έρευνα για την ασφάλεια, έχουμε φτάσει πολύ πιο πέρα από τα πρότυπα που είμαστε διατεθειμένοι να εφαρμόσουμε και πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε θα φροντίσουμε να εφαρμοστούν πολιτικά τα πρότυπα για τα οποία είμαστε βέβαιοι. Ε, την ε, ιδέα να επικεντρωθούμε στον παροπλισμό και ε, στην τελική αποθήκευση των αποβλήτων, αυτή δεν την έβγαλα από το πουθενά. Θα γνωρίζετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στους τομείς αυτούς, όχι μόνο λόγω των αποφάσεων εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας ε, και στη Γερμανία είναι μάλλον μικρότερο το, πρόγραμμα από αλλού, το πρόβλημα από αλλού. Ε, στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι εμπειρογνώμονες λένε ότι υπάρχει η διάθεση ε, να αποσυνδεθούν ε, οι παλαιότερες εγκαταστάσεις, οι παλαιότεροι αντιδραστήρες, αλλά ε, με την χρεοκόπηση της βέβαια η ΕΝΤΕΕΦ δεν έχει καθόλου τους απαρότητους πόρους. Αυτό το θέμα δεν συζητιέται επαρκώς. Τι γίνεται δηλαδή όταν έχουμε κακοδιαχείριση πυρηνικών επιχειρήσεων όταν δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές ε, δεν είναι πια σε θέση να διασφαλίσουν τον παροπλισμό. Και λένε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ε, τα παλιά εργοστάσια ε, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε τα χρήματα για τον παροπλισμό τους. Κύριε Χένκελ, ακριβώς αυτή η περίπτωση, η χρεοκόπηση της Αρίβα, χρεοκοπία της ε, Αρίβα ε, δείχνει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Ε, αν εμπιστεύεστε μόνο τα νούμερα θα δείτε ότι είναι πολύ εντυπωσιακά και με πολύ αρνητικό τρόπο. Υπέβαλα κάποιες προτάσεις. θα έχουμε περαιτέρω συζητήσεις διότι καταλαβαίνω ότι δίστανται οι απόψεις ε, και θα δούμε εάν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία εισηγήτρια. Να σας θυμίσω ότι 26 Απριλίου είναι δηλαδή μεθαύριο το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, ε, ψηφοφορία στην Ήτρε 10 Ιουλίου και Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συναντηθούμε στις 1.30 στο διακοινοβουλευτικό φόρουμ της ενεργειακής κοινότητας. Σας προσκαλώ λοιπόν να συμμετάσχετε ε, στην ε, συνάντηση αυτή με συναδέρφους από εννέα κράτη της ε, Ανατολικής Ευρώπης. Και συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας στη 2.30 σήμερα το απόγευμα. Α, κυρία Χάρμς. Ε, λυπούμε πολύ, δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η συνάντηση αυτή, ε, επειδή θα συμμετάσχουν και συνάδελφοι από την Ανατολική Ευρώπη. Αλλά πρέπει να πάω στο Κίεβο, λόγω της 32ης επαιτίου του Τσερνομπίλ. Ε, θα έχω λοιπόν πράγματα να σκεφτώ τώρα μετά την σημερινή συζήτηση. Και όπως είπαμε, στις, μια, στις μία θα έχουμε γεύμα ε, στο ίδιο μέρος όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τους ε, συναδέλφους. Σας προσκαλώ λοιπόν και σε μεσημερινό γεύμα. Ευχαριστώ. I didn't